στην ημερήσια διάταξη για τις ψηφοφορίες. Έχουμε να ψηφίσουμε 7 προτάσεις ψηφίσματος για την κατάσταση στην Κούβα. Περνάμε λοιπόν στην πρόταση, στην κοινή πρόταση ψηφίσματος 6 πολιτικών ομάδων. Θέλει κάποιος το λόγο. Κύριος Γκόμπερ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να περιμένουμε λίγο ακόμα γιατί μερικοί συνάδελφοι είναι ακόμη στους ανελκυστήρες γιατί κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να κλείσει τους ανελκυστήρες να τους συντηρήσει τη βδομάδα που είναι η σύνοδος γι' αυτό παρακαλώ περιμένετε Ναι κύριε Γκέμπελς Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε περάσει όμως τις 12. Έχει 5 λεπτά που περιμένουμε. Επομένως νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Τροπολογία υπαριθμών 2 της ομάδας της Ηνωμένης Αριστεράς. Ψηφοφορία κατά ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Αφήνουμε λίγο ακόμα ανοιχτό για να ψηφίσω και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10. Ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η παράγραφος 10. Τροπολογία υπαριθμών 1. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Με πολύ μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται το κοινό ψήφισμα, επομένως καταπίπτουν τα υπόλοιπα. Συγχαρητήρια σε όσους εκπώνησαν το κείμενο. Στη συνέχεια έχουμε δύο προτάσεις ψηφίσματος για την επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος τριών πολιτικών ομάδων. Τροπολογία 14. Ψηφοφορία χωρίς ονομαστική κλίση. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 8. Ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία 9. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση την ε, τροπολογία 10. Άρχεται, διορθώνει ο Πρόεδρος τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται η τροπολογία 4. Παράγραφος 14. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Τροπολογία 10 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. ...πέρα της ψηφοφορίας. Η τροπολογία 10 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 5 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία 5. Ψηφίζουμε την τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία 16. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμό 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 17 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Η τροπολογία 19 εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Η 18 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές να επαληθεύσουμε άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέραν της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία 1. Τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Η τροπολογία 2 απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να δούμε ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται η τροπολογία 3. Ψηφίζουμε. Το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Με πριο ψηφία εγκρίνεται το ψήφισμα. Ε, καταπίπτουν τα υπόλοιπα. Συγχαρητήρια. Να περάσουμε τώρα Θέλει κάποιος να παρέμβει? Όχι. Περνάμε τώρα σε πέντε προτάσεις ψηφίσματος για την φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και τις επιπτώσεις από την καταιγίδα Ξύνθια στην Ευρώπη. Περνάμε λοιπόν στην εξέταση της πρότασης ψηφίσματος που υπέβαλαν πέντε πολιτικές ομάδες. δύο τροπολογίες στις παραγράφους 3 και 4. Η ε, τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία 10. Τροπολογία 7 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Η τροπολογία 7 απορρίπτεται. Η τροπολογία 11 αποσύρθηκε. Τροπολογία 8 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato tutti. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Η τροπολογία 8 απορρίπτεται. Τροπολογία 12 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Η τροπολογία 12 απορρίπτεται. τροπολογία 13 υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία να κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. το συγγνώμη. Έκανα λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Όχι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγώ για σας το κάνω επειδή χιονίζει για να τελειώνουμε. Πέρασε ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Καταπίπτουν οι υπόλοιπε προτάσει. Να περάσουμε τώρα στις επεξηγήσει ψήφου. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο Μύροσλαβ Μικολάτσης για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, podľa archívov štátnej správy a dostupnej literatúry Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε.